Good morning. Dear colleagues, good morning. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε πρωί πρωί. Πρέπει, αλλά προηγουμένως πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Συνεπώς, προτείνω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με την εξής αλλαγή. Πρώτον, σημείο 8 που είναι η γνωμοδότηση τη ΛΥΜΠΕ για την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου στο διαζύγιο να αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίασή μας. Δεύτερον, μετά την ψηφοφορία θα συζητήσουμε το σημείο 5. Πρόκειται για τις διαπραγματεύσεις τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία TFTP. Και κλεισμένο το θυρών θα γίνει αυτή η συζήτηση μετά από αίτηση της Επιτρόπου Μάλστρομ, που είναι αρμόδια για τις διαπραγματεύσεις και οποία θα έρθει εδώ να συζητήσει μαζί μας. Συμφωνούμε? Παρακαλώ κύριε Κόγιο. Πρόεδρε. Την τελευταία φορά που συζητήσαμε για αυτό το θέμα, επιτρέψαμε στο Συμβούλιο να είναι παρόν. Γιατί είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο το Συμβούλιο να γνωρίζει τι αποφασίζουμε εμεί. Θα είναι το Συμβούλιο, εντάξει. Α, άμα είναι εδώ και το Συμβούλιο, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ναι, ωραία, συμφωνούμε γι' αυτό. Συνεπώς, Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Πρώτον, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η έκθεση Κάσμαν για την πρόσβαση στα έγγραφα και τη διαφάνεια είναι μια έκθεση για την οποία παρατείνουμε την προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Έχει κυκλοφορήσει βέβαια αυτή η πληροφορία ήδη από τη Δευτέρα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πρέπει να την έχετε πάρει. Έπειτα, ε, μετά από αίτηση της κυρίας Ματιέ, που είναι η συγγήτρια για την ενιαία άδεια, ενώ αρχικά είχαμε προθεσμία 31 Μαΐου, τελικά τώρα είναι 13 Ιουλίου. Αναβάλλεται συνεπώς. Τρίτον, προτείνουμε